Περνάμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Λανσμπέργκης. Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας, μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης. Θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Λανσμπέργκης. Πού είναι? Δεν τον βλέπω. Δεν θέλει προφανώς να πάρει το λόγο. Όχι, νομίζω πως ναι. Πάρα πολύ σύντομα, κύριε. Στο Πρόεδρε, η Γεωργία είναι πολύ προχωρημένη στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τη Συμφωνία Σύνδεση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ο πληθυσμό τη Γεωργία είναι υπέρ τη ευρωπαϊκή πορεία. 68% θέλουν η χώρα του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουν τη δημοκρατική ανάπτυξη τη χώρα. Η εισβάθο και σφαιρική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών έχει θετικέ επιπτώσει στη γεωργία με τι συνεχείς μεταρρυθμίσει. αλλά λόγω τη ασυμμετρίας οι επιπτώσει ε, στο εμπόριο ε, να συμμετρία στο εμπόριο, ε, η ευρωπαϊκή αγορά δεν θα αισθανθεί την επίπτωση. Η Γεωργία όμω κερδίζει σε θέσεις απασχόλησης, ε, αυξάνει τι τις τη, ανάπτυξη και έχει και ένα ε, καλό περιβάλλον για τι επιχειρήσει. Ο προτινόμενος κανονισμός έχει τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπουν την επανεισαγωγή του τελωνιακού δασμολογικού συντελεστή του πλέον ευνοούμενου κράτους. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξετε αυτή την έκθεση. Είναι ενιαία έκθεση με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Περνάμε στην επικύρωση της συνθήκης του Μαρακές βάσει των αναφορών που ελήφθησαν κυρίως τις 9.24 του 2011. Είναι ψήφισμα με ενιαία ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά αποχές υιοθετείται. Περνάμε στη διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106, έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων σόγιας FG72, ε, που την προτείνει η Επιτροπή Υγείας. Τροπολογία 3, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πρώτη τροπολογία. Διανατάσσεω τη χειρό υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψυχοφορίας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα συνολικά με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε το ψήφισμα. Δεύτερο θέμα που αφορά γενετικώ τροποποιημένη σόγια. Ε, πρόταση ψηφίσματος ίδιας επιτροπής. ΜΟΝ 87 και ΜΟΝ 89788. Τροπολογία 3 ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε. Διαντάσσος χειρός στην τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία την τροπολογία 2. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το, το ψήφισμα συνολικά με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε το ψήφισμα. Τρίτο ντοσιέ του ίδιου στυλ για την ε, γενετικά τροποποιημένη σόγια. Τροπολογία 3. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Πρόκειται για το μόνο και μόνο 89-788. Πέρα ψηφοφορίε. Απορρίπτεται. Δυνατά ισχυρό. Ψηφίζουμε την τροπολογία. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία του ψηφίσματος συνολικά. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από λεφρά επιβατικά και εμπορικά οχήματα. Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος ε, προτείνει αυτό το ψήφισμα. Η κυρία Βιένκοβα νομίζω θέλει να πάρει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Παρακαλώ ησυχία, συναδελφοί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Θα διαβάσω μια επίσημη δήλωση της Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να τονίσω πριν ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν κοινό συμφέρον. Την τελευταία εβδομάδα μπορέσαμε να παρουσιάσουμε ε, ένα στεναρό σύστημα στην Ευρώπη. Θα έχουμε ως Κομισιόν ε, εποπτικές ε, αρμοδιότητες και τα κράτη-μέλη θα εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουν τους κανόνες. Τώρα θα ήθελα να περάσω στην επίσημη δήλωση της Κομισιόν. Η Κομισιόν δεσμεύεται να υιοθετήσει διαδικασία δοκιμών από το Σεπτέμβριο του 2017 για να μετρήσουμε τις πραγματικές εκπομπές συνθήκες οδήγηση ε, βασιζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην υποστήριξή του προς αυτήν την κατεύθυνση. Τον Οκτώβριο, στις 28 Οκτωβρίου του 2015, η Επιτροπή ε, ψήφισε ένα ε, κανονισμό της Κομισιόν για τα όρια στα επιβατικά, ελαφρά επιβατικά οχήματα. Ξέρουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα της προφορίας ε, στη TCMV ε, οδήγησε σε κριτικές ε, από το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τον παράγοντα συμμόρφωση. Πιστεύουμε ότι ο μηχανισμό αναθεώρηση του σχεδίου κανονισμού είναι το κατάλληλο εργαλείο για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι κριτικέ. Η ετήσια έκθεση για τον δεύτερο παράγοντα συμμόρφωση υπάρχει ρητά στο σχέδιο κανονισμού τη Κομισιόν. Η αντίρρηση ε, αυτή τη ρήτρα αναθεώρηση είναι ο παράγοντα συμμόρφωση να φτάσει στο 1 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2023 η Κομισιόν δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει αυτή τη ρήτρα αναθεώρησης για να μειώσει ε, το δεύτερο παράγοντα συμμόρφωσης το 2017 ήδη και σε αιτήσια βάση. Λόγω της ρήτρας αναθεώρησης και των τεχνικών βελτιώσεων που αναμένουμε, οι κατασκευαστές από σήμερα θα πρέπει να σχεδιάζουν αυτοκίνητα τα οποία συμμόρφονται με παράγοντα συμμόρφωσης 1. Η Κομισιόν καλωσορίζει την έκθεση αυτή την έκθεση για το θέμα αυτό και συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη να εξασφαλίσει ότι η Κομισιόν έχει τις αρμοδιότητες να υφετεί μέτρα για τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και για τους παράγοντες συμμόρφωσης μέσω εκτελεστικών ε, συμπράξεων. Η Κομισιόν θα συνεργαστεί πιο στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να φτάσει σε συμβιβασμό με αυτό το σκοπό και μάλιστα μελητή η Κομισιόν ούτως ή άλλως θα εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εμπλέκεται όπως πρέπει σε ό,τι αφορά τα θέματα του παράγοντα συμμόρφωσης ε, του δεύτερου. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία των δύο συνομοθετών θα μας επιτρέψει ένα νέο αποτελεσματικό αξιόπιστο πλαίσιο έγκρισης για τα επιβατηγά οχήματα. Ευχαριστώ και το πλήρες κείμενο της δήλωσης Κομισιόν θα σας δοθεί σε εσά και στις υπηρεσίες σας. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ΕΜΔΙΟ, ο κύριος Λαβία, παίρνει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μπιανκόφσκα για την παρουσία της σήμερα στην Ολομέλεια και τον Αντιπρόεδρο κ. Σεύκοβιτς για την σημαντική δουλειά που κατέβαλαν. Η δήλωση είναι απόδειξη θετικής διοργανικής συνεργασίας και αποτελεί σαφή δέσμευση για το μέλλον καλώ όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβουν υπόψη αυτή τη δέσμευση κατά τη διάρκεια της ε, ψηφοφορίας που είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του ψηφίσματος συνολικά. Χρειάζεται ειδική πλειοψηφία και θα γίνει ονομαστικά η ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. Δεν χρειάζεται, απαιτείται ε, ειδική πλειοψηφία 375 μελών δεν επιτεύχθηκε. Άρα απορρίπτεται το ψήφισμα. Έκθεση Reading. Διαπραγματεύσεις επί της Συμφωνίας για τις συναλλαγές του τομέα των υπηρεσιών. Τη Επιτροπή διεθνού εμποδίου. Τροπολογία 64. δυνατά των χειρών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66. Πάλι ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. διανατάσεις των χειρών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστικά. Η τροπολογία 22 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23 τροπολογία διανατάσεως 23 διοθώνει πρόεδρος 23 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ονομαστικά ή τροπολογίες 325 ταυτόσιμες άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 26 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρα τη Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 4. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Παράγραφος 1. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές δεν κατάλαβα τίποτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με ονομαστική ψηφοφορία 65 άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 29 ονομαστικά πάλι. Πέρας, ε, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 με διαναστάσεις υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος ονομαστική ψηφοφορία για το 5. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρασε δύο ψήφοι. Ήταν στο τσακ πάντως. Παράγραφος 1 B, V. Το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρα κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το απολογέ 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το 31 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται με ονομαστική ψηφοφορία η 54 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται παράγραφος 1 σε 9 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, μόνο τα υπέρ είδα. Εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί σταματάτε να σηκώνετε τα χέρια σας. Δεύτερο τμήμα. Αρχικό κείμενο. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Να σηκώνει το χέρι σας συνάδελφοι. Τροπολογία 36. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Διονομαστικής ψηφοφορίας η τροπολογία 37 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1D5. Διανατάσεις των χειρών ψηφίζουμε το κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το 38 απολογεί, ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. απολογεί 39 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Διονομαστικής ψηφοφορίας η 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ονομαστικά η 42. υπέρα. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 43 διανατάσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστικά η 44 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 45 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 46 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας Αποδείπτεται. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1Ζ9. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Διανατάσεως. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά θα ήθελα να το ελέγξουμε 49 ψήφος επαλήθευσης ψηφοφορία επαλήθευσης πέρας απορρίπτεται 50 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 51 διανατάσεως υπέρ. Κατά. Απχές. Απορρίπτεται. 53 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 με ανατασχυρών Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 διανατάσεως. Μάλλον εγκρίνεται και από εκπίπτει. 68 με ονομαστική κλίση. Πέρας. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 διανατάσεως. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. 9. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Διανατάσεως. Άρχεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 με κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 δε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ονομαστική κλίση για την 1 η άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη νέα στατηγική για ισότητα ανδρών και γυναικών και τα δικαιώματα των γυναικών μετά το 2015. Πρόταση ψηφίσματος της ομάδας EFDD. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται κοινό ψήφισμα σοσιαλιστών, φιλελευθέρων, γκουε και πρασίνων. Παράγραφος 1. Αρχικό κείμενο μονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2 με ονομαστική κλίση και πάλι το αρχικό κείμενο άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2D με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 με ανάταση χειρών υπέρ κατά αποχές να κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό για την 10. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές να κάνουμε επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της 12 άρχεται πέρας απορρίπτεται εκπίπτει το δεύτερο τμήμα κατά συνέπεια τροπολογία 11 σε δύο τμήματα επίσης πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό Πρώτο, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 11 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απολύτως τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 15, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 15 δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Ναι, ναι. Ήταν πολύ μικρή διαφορά, αλλά απερίφθη. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράφος 4 σε δύο τμήματα. Το αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα. Συγγνώμη, η 16. Έλεγχος 16. Ηλεκτρονικός έλεγχος για 16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράφος 4. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήματα υπέρ. Αποχέ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο εκπίπτει, περνάμε στην τροπολογία 5 μονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, σε ελέγξουμε όμως. 14 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 6 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 7D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Προς το απορρίπτεται αλλά ας κάνουμε ηλεκτρον... Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ονομαστική κλίση στο νοτιολογική σκέψη α αρχικό κείμενο άρχεται πέρας εγκρίνεται 9D ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη σίγμα τάφ. Αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κλείνουμε λοιπόν την, ε, ψηφοφο... την, ε, τις ψηφοφορίες και διακόπτεται η σύνοδος. Les αρχίσουν τώρα οι επεξηγήσεις ψήφου.